Ξεκινήσουμε με τι ανακοινώσει στα γερμανικά. Οι αρμόδιε Ισπανικέ Αρχέ με ενημέρωσαν για την έκλογη του κ. Λικιάν Καλτσαμπών από 20 Νοεμβρίου 2018. Ο κ. Καλτσαμπών αντικαθιστά τον κ. Σουνξαβάγκα. Οι αρμόδιε Βουλγαρικέ Αρχέ με ενημέρωσαν για την εκλογή του κ. Ανδρέ Νοβακόφ από 24 Νοεμβρίου 2014. Ο κ. Νόβακοφ αντικαθιστά τον κ. Ντόντσεφ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημειώνει την εκλογή του κ. Κολτσαμπών και του κ. Νοβακόφ από την εκάστοτε ημερομηνία έναρξη, από, σύμφωνα με το άρθρο 7, σε ό,τι αφορά τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού. Καλώς ορίζω τους νέους συναδέλφους. Να υπενθυμίσω ότι σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 του κανονισμού, έχουν πλήρη δικαιώματα και με πλήρη δικαιώματα μπορούν να συμμετέχουν στις ε, συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των οργάνων τους όσο δεν έχει ελεγχθεί η εντολή τους ή δεν έχει αμφισβητηθεί η εντολή τους και υπό τον όρο ότι ε, θα δηλώσουν εκ των προτέρων ότι δεν κατέχουν οποιαδήποτε θέση η οποία δεν συνάδει με την εκτέλεση θητείας ως Ευρωβουλευτού μία δεύτερη παρατηρήση, μία δεύτερη ανακοίνωση και μία τρίτη. Σύμφωνα με τα του κώδικα δεοντολογίας στις 25 Νοεμβρίου 2014 αποφασιστικά τώρα του Τζον Μαρί Καβαντά ως μέλο της Συμβουλευτικής Επιτροπής ε, για την συμπεριφορά